Τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω ένα, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Αντιπρόεδρο, συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μογκερίνη. Περνάμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Είναι μια δήλωση της κυρίας Μογκερίνη για την κατάσταση στην δημοκρατία του Κογκό. Εφόσον είστε έτοιμοι μπορείτε να πάρετε το λόγο, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων την οποία αποφασίσατε να οργανώσετε σήμερα για την Δημοκρατία του Κόγκο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως γνωρίζετε είναι εταίρος, ισχυρός και διαρκής της χώρας αυτής τα τελευταία 15 χρόνια. Από το 2006 εμείς ε, στηρίξαμε και οργανώσαμε οικονομικά τις πρώτες ε, ε, ελεύθερες εκλογές και ενισχύουμε γενικά την χώρα αυτή. Έχουμε κάνει δύο στρατιωτικές παρεμβάσεις, έχουμε κάνει επίσης και δύο αποστολές στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και έχουμε βοηθήσει και σε τομείς όπως η διαχείριση των φυσικών πόρων. Σήμερα πολλοί από εμά ανησυχούν για τις καθυστερήσεις γύρω από την επερχόμενη εκλογική διαδικασία η οποία προβλέπεται ε, να γίνουν οι εκλογές το 2015 ε, προεδρικές και 16 βουλευτικές το αργότερο. Ε, οι τελευταίες εκλογικές ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει λαϊκές αντιδράσεις με πάρα πολλά θύματα οι στιγμές είναι δύσκολες και γι' αυτό ζητάμε από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αναζητήσουν ε, την συνένεση να γαλινέψει η κατάσταση και ζητάμε από την κυβέρνηση να κρατήσει τον χώρο της πολιτικής διαβούλευσης ανοιχτό. Προϋπόθεση, ε, η προϋπόθεση της οργάνωσης μιας γενικής απογραφής δεν ισχύει πλέον και αυτό δίνει την δυνατότητα να οργανωθούν οι εκλογές στα πλαίσια του προβλεπόμενου από τον συνταγματικό χάρτη της χώρας ε, χρονικού πλαισίου. Είναι κάτι το οποίο καλωσορίζω και ελπίζω και πολλοί να στηρίξουν τη διαδικασία αυτή. Ε, έτσι και αλλιώς ο σεβασμός του συντάγματος είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι ο απλός σεβασμός μιας συγκεκριμένης ρύθμισης για τις χρονικές προθεσμίες. Ο σεβασμός επίσης των απόψεων της αντιπολίτευσης είναι κριτήρια για την αξιολόγηση της δημοκρατίας στην χώρα αυτή. Πρέπει εμείς να είμαστε σε διάλογο λοιπόν με την κυβέρνηση αυτής της χώρας και να τους πείσουμε να μειώσουν την ένταση στο εσωτερικό επίπεδο. Σημερίζομαι τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το νοσοκομείο Πάντζη και τον, δόκτορα, τον δόκτορα Μουκουέγκα και εγώ είχα ακούσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα τα δραματικά του λόγια τον προηγούμενο Νοέμβριο στα πλαίσια της απονομής του βραβείου Σαχάροφ και είχα τη δυνατότητα ε, να τον συναντήσω, να ανταλλάξουμε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις ε, σχετικά με την βοήθεια προς τη χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την φυσική ασφάλεια του ιατρού ε, στα πλαίσια της προσπάθειάς του ε, σαν προσπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζήτησα επίσης ε, στην σας από τον αντιπρόσωπό μας να διαμεσολαβήσει στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και στο, νοσοκομείο Πάντσι. Νομίζω ότι η μετάβαση στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών έχει μεγάλη σημασία για τη σταθερότητα όχι μόνο στη χώρα αυτή αλλά στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε να εξουδετερωθούν όλες οι ένοπλες ομάδες στην ανατολική πλευρά της χώρας χάρη στις προσπάθειες της Μανούσκο και, της, του οργανωμένου στρατού έχει υπάρξει πρόοδος οι κυβερνήσεις της Ρουάντα, της Ουγκάντα και ε, του Κονγκό θα πρέπει να συνεννοηθούν για να οδηγήσουν στον αφοπλισμό αυτών των ένοπλων ομάδων. Υπάρχει μια ομάδα βέβαια ένοπλη η οποία εξακολουθεί να απειλεί τη χώρα. Συνδέεται ε, και με την ιδεολογία της γενοκτονίας της Ρουάντα στο παρελθόν έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα. Η υποστήριξη λοιπόν των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε στην περιοχή αυτή τις αιτίες της σύγκρουσης. Το κίνημα αυτό είχε χρόνο έτσι ώστε να οργανώσει ειρηνικά την παράδοσή του. Το συζητήσαμε αυτά την προηγούμενο Ιανουάριο, ε, τον Ιανουάριο που πέρασε και καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Είπαμε ότι έχει έλθει πλέον η στιγμή για να οργανωθεί μια στρατιωτική παρέμβαση εναντίον αυτών των ομάδων. Ζητήσαμε επίσης από τη Μονούσκο και από τον στρατό να προστατεύσουν τους, ε, ε, τους ε, αμάχους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι στηρίζουμε την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. Στηρίζουμε τις προσπάθειες και της Μανούσκο και όλων των στρατιωτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν, όπως επίσης και τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών. Να υπογραμμίσω, Πρόεδρε, ότι και εμείς συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για τη διασύνδεση τη σύγκρουση της ένοπλης από τη μία με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από την άλλη. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε, και ή προκατοχός μου είχε κάνει μια επίσημη ανακοίνωση για το πρόβλημα των, των που προέρχονται από παράνομα κατεχόμενες περιοχές. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν σαφέστατες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από πλευράς μας για την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και των εθνικών πάρκων μεταξύ των οποίων και του πάρκου Βιρούγκα που απειλείται από αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων για ανείχνευση ε, ποσοτήτων πετρελαίου στην περιοχή. Εμείς θα ελέγξουμε τις εθνικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την αηφόρο επιβίωση του συγκεκριμένου φυσικού πάρκου. Ε, ζήτησα από τον κύριο Φερβέκε, τον υπεύθυνο για τις μεγάλες λίμνες, αποκινούμε τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών να πάμε στην Κινσάσα για να αξιολογήσουμε επιτόπου την περιοχή για μια ακόμη φορά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα ακούσω με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και τώρα ξεκινά η συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριο Στυλ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει διάφορα προβλήματα. Η ύπατη πρόσωπος έχει αναφέρει κάποια από αυτά όπως ας πούμε η παράνομη χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων, την συστηματικό βιασμό των γυναικών για τον οποίο ε, αναφέρθηκε, μίλησε εδώ ο Δόκτωρ Μακουέγκα κλείσε και το νοσοκομείο του δόκτωρος Μακουέμπα αφού επέκρινε τις αρχές. Τα αίτια όλων αυτών των προβλημάτων όμως βρίσκονται στις μη αποτελεσματικούς δεσμούς, τους μη δημοκρατικούς θεσμούς, την έλλειψη ένομης τάξης και του υψηλού επίπεδου διαφθοράς. Αυτοί που διαμαρτύρονται στην ε, Κινσάσα εξεγέρθηκαν γιατί πρόκειτο να αλλάξει ο εκλογικό νόμος εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ήταν απόλυτα σαφές ότι η, αλλαγή του εκλογικού νόμου ήταν προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία ο πρόεδρος Καμπίλα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο εκδημοκρατισμός και η διαδικασία της πρόθεσης της δημοκρατίας στη χώρα, όπως επίσης να υπάρξει συνεργασία για την ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν δημοκρατικοί θεσμοί ε, για όλους. Πιστεύουμε ότι ότι αυτό αφορά και την αναπτυξιακή πολιτική αλλά και την γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι αυτό ένα ξεκάθαρο μήνυμα ε, του ε, Κοινοβουλίου. Παρότι σήμερα υπάρχει μια ε, κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Καμπίλα και προηγουμένως του πατέρα του, η οποία είναι κυβέρνηση ε, μη δημοκρατικοί ε, ε, πιστεύουμε ότι μπορούν να αλλάξουν τα, οι θεσμοί. θα ήθελα να πω ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην αποκατάσταση της δημοκρατίας αλλά και τη σταθερότητα γενικά των χωρών των μεγάλων λιμνών, της περιοχής των μεγάλων λιμνών. Φοβάμαι ότι λαμβάνονται μέτρα τα οποία απομακρύνουν τους πολίτες από τη δημοκρατία. Η σωστή διακυβέρνηση και η εναλλαγή στην εξουσία είναι κάτι που λείπει από τις περιοχές αυτές. Υπάρχουν χιλιάδες νεκροί μόνο και μόνο γιατί διαμαρτυρήθηκαν πολύ ε, νόμιμα εναντίον της τροποποίησης του εκλογικού νόμου. Καταδικάζουμε τη σύλληψη του Κιβόκο και άλλων προσωπικότητων της τοπικής αντιπολίτευσης και ζητάμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Καταδικάζουμε τη βία εις βάρος των γυναικών. Οι τρομερές αυτές ενέργειες πρέπει να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Πρόεδρε, πρέπει να γνωρίζει κανείς την αξιοπρέπεια του αντιπάλου στα πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Έτσι μόνο θα αποφύγουμε τη βία και έτσι θα πρέπει να δράσουν και οι ομάδες οι πολιτικές στο Κονγκό. Καμία παραβίαση όμως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα γίνει ανεκτή από την διεθνή κοινότητα και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Γι' αυτό λοιπόν θα υποστηρίξουμε την απαστολή Μονούσκο στο σύνολο του εδάφους του Κονγκό. Και τέλος, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι ντρέπομαι σαν Ευρωπαία πολίτης για μία ακόμα τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 29 παράνομους μετανάστες κοντά στη Λαμπεντούσα. Άνδρες, γυναίκες, παιδάκια που απλά ήταν ένοχοι γιατί ήθελαν μια καλύτερη ζωή. Ο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, θέλω να συγχαρώ και εγώ την είπατε εκπρόσωπο για την εξαιρετικά σαφή και συγκεκριμένη σύνοψη που έκανε που δείχνει την δέσμευσή μας απέναντι στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό η οποία ε, εκρήγνεται πράγμα που έχει επιπτώσει και στην ευρύτερη ε, περιοχή. Πρέπει η Προεδρία να είναι... Ε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προθεσμίες και να δούμε ανάλογα με αυτές. Ο κύριος Βιαμανουβαλού πρέπει να μην καθυστερεί. Αυτή είναι απέτηση της διεθνούς να, της διεθνούς κοινότητας να μην καθυστερεί να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα. Θέλω να ε, χαιρετήσω τον πρόεδρο της Γερουσίας ε, που είχε το θάρρος να ε, αρνηθεί το άρθρο 8 το οποίο θα καθυστερούσε τουλάχιστον επί τρία χρόνια την, ε, τις εκλογές και θα πρέπει οι εκλογές να γίνουν σε κλίμα ήρεμο χωρίς βία ε, κατά της κοινωνίας των πολιτών, των πιθανών υποψηφίων και των δημοσιογράφων. Η ελευθερία του τύπου, της έκφρασης και της ειρηνικής διαδήλωσης είναι θεμελιώδη δικαιώματα που, πρέπει, που τα εγγυώνται το Σύνταγμα και επιμένουμε σήμερα επ' αυτού ε, τώρα. το γεγονός ότι ε, ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν επιθέσεις κατά των ε, δυνάμεων απελευθέρωσης της Ρουάντα είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Ξέρουμε ότι αυτά τα θέματα που, της γενοκτονίας που δεν έχουν επιληθεί αποτελεί, αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η προστασία του άμαχου πληθυσμού της περιοχής, των γυναικών και των κοριτσιών που πέφτουν θύματα άνθρωπων πράξεων και επαναλαμβάνω την εξαιρετική εργασία που έκανε ο τιμηθής με το γραφείο ε, Ζαχάροφ γιατρός και, και παρά το ότι τιμήθηκε με το βραφείο ε, έχει πέσει θύμα εκφοβισμού. Γι' αυτό τον τρόπο θα πρέπει να υποστηρίξουμε ένα είδος παρατηρητηρίου με τα Ηνωμένα Έθνη και τις ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρακολουθούμε την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Επόμενος ομιλητής, η κυρία ε, Σένρα Ροντρίγκες, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να πω ότι κάθε σύγκρουση την οποία αναλύουμε και εξετάζουμε σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο συνδέεται πάρα πολύ συχνά με τα συμφέροντα των μεγάλων πολιεθνικών εταιριών και τα συμφέροντα των δυτικών δυνάμεων στην εκμετάλλευση για να μην πω λάτιση των φυσικών πόρων των συγκεκριμένων χωρών. Στην περίπτωση της Δημοκρατίας του Κογκό δεν μας διαφεύγει η τεράστια στρατηγική σημασία που έχει λόγω του τεράστιου γεωγραφικού του μέγεθους. Η χώρα αυτή έχει τεράστιες ε, φυσικές πηγές, πετρέλαιο, ουράνιο, διαμάντια κτλ. Είναι μια χώρα πάμπλουτη και ταυτόχρονα μια χώρα πάμπτωχη. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση στις συγκρούσεις αυτές. Θα πρέπει ε, να δούμε τι πρέπει να γίνει με τις πολυεθνικές, πρέπει να φύγουν από αυτές τις χώρες και θα πρέπει οι ίδιοι οι κάτοικοι να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους και να κερδίσουν από την οικονομία της χώρας τους και θα πρέπει να προστατεύουμε τις γυναίκες και τα παιδιά γιατί είναι τα πρώτα θύματα τέτοιου είδους καταστάσεων. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαμπζεντίνη, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα ακόμα χρόνο πριν από τις εκλογές και βλέπουμε ότι κλείνει το Facebook, υπάρχουν όλο και πιο μεγάλες επιθέσεις, οι ακτιβιστές απειλούνται. Και το τονίζω αυτό ότι μένει ένας χρόνος μέχρι τις εκλογές, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε να μην καθυστερήσουν οι εκλογές και η δύο θητεία για το Καμπύλε να μην είναι δύο θητείες. Να το τονίσουμε αυτό. Να προσέξουμε λοιπόν το τι συμβαίνει στο Κονγκό με τους ακτιβιστές που χρειάζονται προστασία. Αλλά πρέπει επίσης να δώσουμε πιο έντονη διαμόρφωση, να διαμορφώσουμε πιο αυστηρά τους στην νομοθεσία μας για τα ορεκτά. Αυτό που ήθελε το Κοινοβούλιο είναι δεσμευτική νομοθεσία για όλα τα προϊόντα που θα οδηγούσε σε βιώσιμη εξόρυξη τέτοιων ορεκτών σε τέτοιε εμπόλεμες περιοχές. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο βγάζοντας τα χρήματα από τον πόλεμο. Πώς θα καθοστήσουμε λοιπόν την ομοθεσία αυτή στεναρή, κυρία Μαγκερίνη. Είμαστε κάπως καθυστερημένοι, λέει η Πρόεδρος, γι' αυτό δεν θα δέχτω μπλε κάρτες. Συζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Κάρβερ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το, η, το Κονγκό είναι ένα κλασικό παράδειγμα δυτικών πολιτικών και το πώς συμπεριφέρονται στα αφρικανικά κράτη σε διπλωματικό επίπεδο. Τα σημερινά προβλήματα είναι άμεση συνέπεια του ψυχρού πολέμου και των, ε, της πολιτικής του βασιλέου του του Δεύτερου που χρησιμοποίησε ως προσωπικό του τσιφλίκι τη χώρα. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ υπό αφρικανική ηγεσία θα πρέπει σήμερα να αποφύγουν να αντιμετωπίσουν τα ερωτήματα, τα ζητήματα που ανακύπτουν από την προηγούμενη συμπεριφορά του σε ό,τι αφορά τι αιτιάσει για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στρατηγό Μαντίβου είναι ακόμα μάχημο κατά, του FDLR. Μπορεί κάποιος που αντιμετωπίζει τέτοιε κατηγορίε να βρίσκεται σε μια τέτοια θέση ισχύω. πώ θα ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο ελπίδα σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαμπριέλ για 1,5 λεπτό λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Εγώ σέβομαι την δημοκρατία του Κονγκό, αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή αυτή της χώρας δεν είναι καθόλου καλή. Η απόφαση της 25ης Ιανουαρίου για τον εκλογικό νόμο δεν θα αποκαταστήσει το κλίμα εμπιστοσύνης. Υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία εδώ. Πρώτον, η δημοσίευση ενός πλήρους χρονικού θα έλεγα προγράμματος για τις εκλογικές διαδικασίες που έτσι και αλλιώς έχει ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή. Μετά από 8 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα. Η κυβέρνηση και οι ΣΕΝΗ δεν μπορεί να συνεχίσουν να κολυσιεργούν. Δεύτερον, το βασικό στοιχείο της εκλογικής διαδικασίας είναι ο διάλογος ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να τον εθωρύνουμε και στα πλαίσια της ομάδας εργασίας της ΣΕΝΗ ή μέσω νέων πρωτοβουλειών που δημιουργούν φόρουμ συζήτησης για την αποκατάσταση με εμπιστοσύνη. Τρίτο μήνυμα. Η εφαρμογή του απόφασης πλαισίου της Άντης. Ε, οι στρατιωτικές δράσεις εναντίον του FDLR δεν μπορεί να είναι αποφασιστικές παρά μόνο εφόσον εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή από όλους. Τέλος, η συζήτηση αυτή ε, μας οδηγεί και στον δόκτορα Μουκβέγγε. Οι αρχές του Κονγκό θα πρέπει να στηρίξουν τη δραστηριότητα του νοσοκομείου του Τάντσι ε, και θα πρέπει επίσης να προστατεύουμε και τις, τους αμάχους ιδιαίτερα από πλευράς του κρατικού στρατού και από την Μονούσκο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αρένα, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο Λουί Μισελ και για το θέμα της ελευθερίας του τύπου και για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για το χρονοδιάγραμμα, το εκλογικό και να υποστηρίξω την πρόταση για το παρατηρητήριο την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως να μην ξεχνά ότι έχει και άλλα μέσα για την άσκηση της πολιτικής της και εννοώ το διεθνές εμπόριο. Συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή Ίντα τα θέματα της καταπολέμησης των λεγόμενων ορυκτών του αίματος Ξέρετε ότι τα θέματα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν στο να πάρουμε μέτρα πίεσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι θα έλεγα ιδιαίτερα συνισταλμένη. Απαιτείται να θυμόμαστε αυτά τα οποία μας είπε ο βραβευμένος από το βραβείο Σαχάροφ δόκτωρας Μουκουέγε που μας ζήτησε να είμαστε θαραλέοι, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και όχι μόνο να καταδικάζουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των υστέρων. Mr. ευχαριστώ. Και εγώ θα υποστηρίξω τις προτάσεις, τις πολύ λογικές, τις οποίες έκανε ο κύριος Μισελ και θα συνενέσω με αυτά τα οποία είπε και η κυρία Ρενά. Εμείς είχαμε συναντήσει πριν λίγο καιρό τον δόκτωρα Μουκέγκουε πραγματικά έχει αφιερώσει τη ζωή τους στις γυναίκες και στα παιδιά ε, που είναι αντικείμενο επίθεσης από όλε τις πλευρές σήμερα. Ο δόκτωρ Μακουέγκε μας ε, ζήτησε να μην αφήσουμε να εκπνεύσει η συμφωνία πλαίσιο της Άντης. Αυτό θα ήταν απαράδεκτο για τη χώρα αυτή και την ευρύτερη περιοχή. Εμείς εμένουμε στις εκλογές το 2015 και το 2016 και ακούγοντας τον δόκτωρα Μουέγκε θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι περνάει από το χέρι μας για να μην υπάρξει ατιμορρησία και να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζοντας όπως είπα τις προτάσεις του κυρίου Λουι Μισελ. Η κυρία Βαλενθιάνο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ είμαι υπέρ της ε, βοήθειας προς τη χώρα αυτή. Μίλησα πριν λίγες ώρες με τον δόκτωρα Μουέγκε και μου ζήτησε να παρέμβει και το κοινοβούλιο μας. Απαιτεί προστασία. Από τις 18 Νοεμβρίου η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Υφίσταται τεράστιες απειλές, εκβιασμούς ε, και μέσω τηλεφώνου και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οι απειλές εις βάρος του προσώπου του και του νοσοκομείου του είναι τεράστιες. Να μην ξεχνάμε τι μας είπε όταν πήρε το φραβείο Σαχάροφ. Μείνανε πάντα τα λόγια του στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση και να πάρει μέτρα ε, δεσμευτικά. Δεν μπορούμε να δίνουμε το Φαβίο Σαχάροφ και να τον αφήνουμε να απειλείται με τέτοιο τρόπο αυτός και οι ασθενείς του. Είναι απαράδεκτη η στάση μας. Και υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη βία την οποία υφίστανται όλων των μορφών δυστυχώς ακόμα και τα παιδιά, όχι μόνο οι γυναίκες. Και γι' αυτό ο δόκτωρ Μουκουέγκε απαιτεί μια διεθνή έρευνα γύρω από την υπόθεση αυτή με άμεση εμπλοκή των ευρωπαϊκών αρχών για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου στην περιοχή αυτή και δίδοντας επαναλαμβάνω εγγυήσει για την ασφάλεια την προσωπική του δόκτωρα Μουκουέγε. Thank you, uh, Mr. Guerrero. Σας ευχαριστώ, κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Μογκερίνη. Η καταστολή της ε, κυβέρνησης της Κινσάσα οδήγησε πριν λίγες μέρες το θάνατο 42 πολιτών. Είναι ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τις χιλιάδες των νεκρών και τις χιλιάδες των εκτοπισμένων, πάνω από 2,5 εκατομμύρια, που ζητούν βοήθεια και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων στους στη χώρα αυτή. Σε αυτό έχουμε καταλήξει και μέσω της δίωξης και εκδίωξης των αρχηγών της αντιπολίτευσης, της δίωξης εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών σε όλες τις μορφές εκπροσώπησής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Αφρικανικής Ενότητας και να εμπλέξει όλες τις πλευρές σε μια ειρηνευτική διαδικασία, σε μια διαδικασία διοργάνωσης ελευθέρων και δημοκρατικών εκλογών. Και τέλος, θα πρέπει να έχουμε μια σαφέστατη πολιτική θέση, ξεκάθαρη πολιτική θέση για την απαγόρευση εμπορίας των παράνομων προϊόντων εξορίξεων στην περιοχή. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να εφαρμόσει αυτά τα οποία είπε η ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Φοντσούλητσα. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Τα πρόσφατα περιστατικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι απαράδεκτα και η εξέγερση της βίας θα πρέπει να καταδικαστεί με όλα τα μέσα. Το Κοινοβούλιο έλαβε μία σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νόμου. Αναμένουμε να θέσει το Κονγκό ημερομηνία για τις προεδρικές εκλογές το 2006. Η ανθρωπιστική κρίση στο Κονγκό επιδεινώνεται κάθε χρόνο, κάθε μέρα με μεγαλύτερες συγκρούσεις για τα ορυκτά, τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλο, τα μέτρα καταστόλης από την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι η χώρα σταδιακά κυλάει στο χάος. Πιστεύω ότι η απειλή των πολιτικών αντιπάλων, των ακτιβιστών θα πρέπει να σταματήσει με κάθε τρόπο και αναμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τα σταματήσει. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για την ασφάλεια του βραβευμένου με το βραβείο Ζαχάροφ ε, δόκτωρας Μουμπέγκεξ που το νοσοκομείο του μπήκε στο στόχαστρο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του εδώ. Θέλουμε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και κόβει πρόεδρο δυστυχώ το μικρόφωνο. Ο πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε, συνάδελφε Φροντζούλικα. Και τώρα περνάμε στη δικασία Catch Το λόγο έχει και ο κ. Μαγιά. κύριε πρόεδρε οι τελευταίες εξελίξεις στη λαϊκή δημοκρατία του κονγκό προκαλούν έντονο προβληματισμό στη διεθνή κοινότητα καθώς η περιοχή αυτή κινδυνεύει με πλήρη αποσταθεροποίηση. αυτό σημαίνει πέραν των άλλων ότι πρέπει να τηρηθούν όσα προβλέπει το σύνταγμα για τη διενέργεια των προεδρικών εκλογών οι οποίες προβλέπονται σε πολύ συγκεκριμένη ημερομηνία. όμως η απόφαση του καμπιλά να επεκτείνει τη θητεία του στον προεδρικό θόκο έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων της αντιπολίτευσης τεράστιες διαδηλώσεις και αιματηρές ταραχές. πολλοί ακτιβιστές έχουν πέσει πλέον νεκροί. η ύπαρξη στρατιωτικών ομάδων και οι τοπικές συγκρούσεις στον κονγκό έχουν όμως ένα υλικό αντικείμενο τον έλεγχο της εκμετάλλευσης των πλούσιων φυσικών πόρων του κονγκό. για τον λόγο αυτό πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να γίνει αξιοποίηση των φυσικών πόρων του κογκό υπέρ του ίδιου του λαού της χώρας. μόνο έτσι θα μπορέσουν να προστατευτούν οι γυναίκες και τα παιδιά στην περιοχή. σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μαριά. Αυτή τη φορά έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ατόμων που έχουν ζητήσει το λόγο όσο και χρόνο ε, έχουμε στην διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τώρα θα δώσω στον συνάδελφο Γευκοφτσής. Η, δημοκρατική, η δημοκρατία του Κονγκό είναι ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη. Όχι επειδή πρόκειται για μια χώρα η οποία ανήκε στον ε, βασιλέα Λεοπόλδο το δεύτερο του Βελγίου στο κονγκό της ε, το σημερινό θέλουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους τους οποίους δικαιούνται οι πολίτες του Κονγκό. Αν δίναμε στον Δόκτωρα Μογκβέγκε, αν δώσαμε στον Δόκτωρα Μογκβέγκε ένα τόσο σημαντικό βραβείο, θα πρέπει και η πολιτική μας να συνάδει με τη βράβευση αυτή. Και γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση προς την ύπατη εκπρόσωπο να επιλύσει την κατάσταση στο Κονγκό με δημοκρατικά μέσα, μέσω των εκλογών, γιατί αυτό θα δείξει ποιος, ε, ποιον, ποιο θέλει ο κόσμος. Σας ευχαριστώ, η επόμενη sur... Θα ήθελα να μιλήσω για την εξορρυκτική δραστηριότητα στη χώρα αυτή. Βλέπετε το κινητό μου κυρία Μογκυρίνη, υπάρχει αίμα σε αυτό το κινητό από τις σπάνιες γέες του Κογκό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο πλουτίζει τις ένοπλες ομάδες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία έτσι ώστε να δρούν με τον τρόπο με τον οποίο δρούν. Έχουμε λοιπόν ευθύνες έχουμε έναν κανονισμό εθελοντικής φύσεως για την προέλευση των ορυκτών, ε, τον ξτένιο, χρυσό κτλ. Θα πρέπει να διευρύνουμε τις ουσίες αυτές και σε άλλους πόρους, ε, να συμπεριλάβουμε το ουράνιο σαν παράδειγμα ή και το πετρέλαιο. Πώς και γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε ο νόμος ε, Dodd Frank να είναι υποχρεωτικός και σε εμά να είναι εθελοντικός. Και δεν θα πρέπει επίσης να υπάρχει ανάγκη πιστοποιητικού μόνο και μόνο για τους εισαγωγείς, αλλά και στον τελικό χρήστη υπάρχει μια δεοντολογία γύρω από την κατασκευή αυτού του τηλεφώνου. Ευχαριστώ κυρία Ριβαζή. Καστάλντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα έλεγε κανείς ότι στη Δημοκρατία του Κονγκό η κατάσταση συνεχίζει να είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είδαμε με τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος προσπάθησε να αναβάλει τις εκλογές. Πάρα πολλές τέτοιες ε, τέος απικίες έχουν ε, πολιτικές τάξεις και ηγεσίε που πιστεύουν ότι η δημοκρατία είναι η δικτατορία η δική τους και όχι η άποψη της πλειοψηφίας του πληθυσμού. Και ο Καμπίλα θέλει να κάνει την χώρα αυτή προσωπική ιδιοκτησία όπως το είχε κάνει κάποτε ο βασιλέας του Βελγίου. Όχι λοιπόν. Εμείς θα πρέπει να μην χρησιμοποιούμε τα βρώμικα αυτά προϊόντα από πρώτες ύλες ματωμένες από τις περιοχές αυτές. Πρέπει τα λόγια του δόκτωρα Μουκουέγκο να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι το βραβείο Σαχάροφ θα είναι το βραβείο της υποκρισίας μας και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Μπονάνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση για το Κογκό βλέπω ότι προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στην Ολομέλεια. Ε, πράγματι νιώθω σαν να βρίσκομαι ε, σε ένα οίκο ευγυρία στην Ιταλία ε, όπου πριν από το βραδινό φαγητό κάνουμε και μια κουβέντα έτσι για να γίνεται. Και πράγματι έτσι όπως μας είπε η κυρία Μογκερίνη μας είπε ότι τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε στο Κονγκό μας παραπέμπει στην Ουκρανία. Πήγε η Μέρκελ να συζητήσει με τον Πούτιν. Ε, νομίζω ότι εσείς δεν είσαστε τίποτα. Είσαστε ένα μηδενικό, είσαστε μια τρίχα για να μην πω κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχετε λοιπόν δεν μετράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν, ορίστε, ξυπνήστε, λέει ο μιλητής, ε, σφυρίζοντας. Κοιμάστε όλοι. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, συνάδελφε Μπονάνο. You have not the floor anymore. Δεν έχετε πλέον το λόγο. Συνάδελφε Μπονάνο. Μιλήσατε και πάρα πολύ και οι τελευταίες σας παρατηρήσεις ε, θα μείνουν εκτός της ε, δημοσιότητας γιατί δεν ε, μπορέσατε, δεν τις μετέφρασαν οι Και έτσι ολοκληρώθηκε η δικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ και δίνει το λόγο στην εκπρόσωπο, στην Αντιπρόεδρο Μογκερίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βλέπω στον κατάλογο των παρεμβάσεων σήμερα το απόγευμα και για τα επόμενα θέματα όπως την κατάσταση στην Ουκρανία και γι' αυτό ο κύριος Μπονάνε δεν είχε ζητήσει να μιλήσει για την Ουκρανία αν θέλει να μείνει εδώ και να πάρει το λόγο. Να πω επίσης ότι πολλοί από εσά αναφερθήκατε σε θέματα τα οποία και εγώ ανέφερα στις προκαταρκτικές μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε τις προσπάθειές μας. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζω ότι το μήνυμά σας είναι ξεκάθαρο και θα γίνει αντιληπτό. Κάποιοι από εσά είπατε ότι αυτό το θέμα δεν είναι μόνο σημαντικό για την ε, χώρα μόνο, αλλά για την περιοχή. Και είναι σημαντικό και για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να δεχθώ την ιδέα ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε τοπικές κρίσεις και σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κοντά στα σύνορά μας. Γιατί αυτό που συμβαίνει και σε χώρες οι οποίες είναι μακριά από τις δικές μας, επηρεάζει την ασφάλειά μας, επηρεάζει γενικότερα τον τρόπο ζωής μας. Δεν είναι μόνο δηλαδή ευθύνη, αλλά είναι συμφέρον ε, της Ευρώπης να είναι πάντα ενήμερο. Να πω επίσης σε κάτι το οποίο μας θύμισε ο δόκτωρ Μουκουέγγε, ο ρόλος των γυναικών. Οι γυναίκες είναι τα μόνιμα θύματα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες, τα κορίτσια, κάθε φορά πιο νέα, κάθε φορά πιο μικρά σε ηλικία, δυστυχώς. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος λοιπόν και ο στόχος αυτός είναι οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι τα πρώτα θύματα αυτής της σύγκρουσης και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι εμείς όχι μόνο εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο στηρίζουμε τα θύματα και σε επίπεδο νομικό και σε επίπεδο ιατρικό, προσπαθούμε επίσης να επηρεάσουμε και κάποιες μεταρρυθμίσεις στον τομέα του δικαστικού σώματος και στον τομέα των δυνάμεων καταστολής. Αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα πιο πολύ με τις γυναίκες που είναι τα πρώτα θύματα όπως είπα σε όλο τον κόσμο. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει ανάγκη εδώ να είμαστε συνεκτικοί με τις θέσεις που είχαμε στο παρελθόν. Όταν δώσαμε λοιπόν το φαβείο Σαχάροφ πριν μερικούς μήνες, αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η υποστήριξή μας δεν είναι προς το πρόσωπο του δόκτωρα Μουκουέγε, αλλά προς τη δουλειά την οποία κάνει και τα επιτεύγματά του. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε εγγυήσει προς το πρόσωπο αυτό και την συλλογική προσπάθεια την οποία κάνει. Γιατί ο δόκτωρ Μουκουέγγε είναι μια ακτίδα ελπίδας για το Κογκό. Για τις προτάσεις του κυρίου Λουί Μισελ. Εγώ κατανοώ το σκεπτικό του, και όταν επανέλθω στις Βρυξέλλες θα μιλήσω με τον κύριο Λαμπρινίδη που είναι ο ειδικό μας εκπρόσωπος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να υποστηρίξουμε την πρότασή του. Ε, επίσης ε, συμφωνώ με τις προτάσεις σας για να ακοπεί ο ομφάλιος λόρος ανάμεσα στα ορυκτά ε, και την ένοπλη βία και αυτά φαίνονται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε την προσωπική μου υποχρέωση. Δεν μπορώ να σας δώσω εγγυήσεις ότι η προσπάθεια θα είναι επαρκής, αλλά η προσπάθεια θα υπάρξει. Τελειώνω ομιλώντας την Ιταλική γλώσσα. Γιατί η κυρία Κέγκε πάρα πολύ σωστά μας θύμισε σήμερα ότι ο θάνατος ξαναγύρισε στη Μεσόγειο χτες. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση και το ότι έθεσε η κυρία Κέγκε το θέμα, να πω ότι μόλις ενημέρωσα το σύνολο των επιτρόπων για την πρόθεσή μου να συγκαλέσω μια έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας των Επιτρόπων για την Εξωτερική Δράση σε συνεργασία με τον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο για να συζητήσουμε πάλι το θέμα της μετανάστευσης να δούμε αν χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα τα οποία έχουμε υπόψη μας και σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο και αναφέρομαι εδώ στις χώρες προέλευσης και τις χώρες διαμετακόμισης και το θέμα αυτό θα το συζητήσει και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Δεν πρέπει να περιμένουμε άλλες τραγωδίες στην θάλασσα. Νομίζω ότι έχουμε τα μέσα, εφόσον έχουμε την πολιτική βούληση, για να αλλάξουμε την κατάσταση. Σας ευχαριστώ, Επιτροπέ Μογερίνη.